Ορθόδοξο Κρεμλίνου. Οπότε έτσι θα πρέπει να αποφασίσουμε να πρέπει να, ε, να επιτρέψουμε να προβεί σε αυτές τις πράξεις το τόσο αμφίβολο καθεστώς του. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Όγιουλάντ. Η σημερινή μας συνεδρίαση ολοκληρώθηκε εδώ. Η αυριανή θα διεξαχθεί αύριο 18 Απριλίου Τετάρτη από τι 9 ω τι 15.00. Η, η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μας και οι εργασίε τη, ε, Εύχομαι σε όλου καλή επιστροφή και καλή ανάπαυση.